witam państwa bardzo serdecznie. και κύριοι μετά τη μεσημεριανή διακοπή αρχίζουμε και πάλι τη συνεδρίασή μας και καλωσορίζω εδώ την Επίτροπο Τάισεν, την προσκεκλημένη μας.